έτσι μπορεί να υπάρξει μια λογική περιφερειακή και διαρθρωτική. Ένα πάγωμα λοιπόν των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και περικοπή τους ακόμα, όπως ε, συζητιέται, μπορεί λοιπόν να ακούγεται έτσι δημοφιλής αλλά θέλω να σας πω εδώ πέρα από τη σκοπιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πως θεωρούμε αυτές τις περικοπές ανεύθυνες. Το να περικόψουμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι θα κόψουμε τον μεγαλύτερο προπολογισμό που προωθεί την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια χρονική στιγμή στην οποία κάποια κράτη-μέλη εξακολουθούν να βρίσκονται σε ύφεση, αυξάνεται η φτώχεια και η ανεργία. Μιλάμε σύμφωνα με τα τελευταία νούμερα για 25,5 εκατομμύρια ανέργων. Οπότε ένα πράγμα χρειάζονται οι άνθρωποι. Δουλειές. Γι' αυτό εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε μια ξεκάθαρη θέση την οποία θέλω να σας αναφέρω. Όχι σε όλα τα σχέδια που θα κάνουν οικονομία μέχρι θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι στην αλληλεγγύη και στι στοχευμένες επενδύσεις στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, την καινοτομία και την έρευνα. Πριν από λίγες μέρε, μαζί με τον πρόεδρο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, βρεθήκαμε σε μια συνάντηση των λεγόμενων φίλων της συνοχής. Εκεί πέρα ήταν 15 από τις 27 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζω πως είναι άρα η πλειοψηφία των κρατών μελών της Και εκεί πέρα συμφωνήσαμε με τις χώρες αυτές το εξής. Η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει και στο μέλλον να παραμείνει κεντρικό στόχος των προσπάθειών μας. Η πολιτική συνοχής είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την άποψή μας για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εμείς δεν θέλουμε μια δογματική προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω με συγκεκριμένα νούμερα και ποσοστά. Αντιθέτως, θέλουμε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, μια ανοιχτή συνολική συζήτηση για το ποιε πολιτικές έχουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Για το πώς λοιπόν θα διαμορφωθεί η μελλοντική πολιτική συνοχής. Ήδη έχουμε κάνει κάποιε διαπιστώσει στο Κοινοβούλιο και διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο. Υπάρχει επίσης μεγάλη αντίσταση στη μακροοικονομική αυτή αίρεσιμότητα μέχρι την εξασφάλιση ενός ποσοστού των διαρθρωτικών ταμείων για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει επίσης να χρηματοδοτηθούν. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες εάν περάσουν την απέτησή τους κάποια κρατημέλη για περικοπή κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Διάσα εφημερίδες το Σαββατοκυριακό και εσείς που αναφέρουν πως μια χώρα θέλει να περικόψει 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα, και σας το λέω εσάς τώρα εδώ πέρα γιατί πρέπει να το ξέρετε, σημαίνει λιγότερα λεφτά για τις περιφέρειές σας, για εσάς, λιγότερη ανάπτυξη της υπαίθρου σημαίνει λιγότερους φοιτητές στο Εράσμους. Σημαίνει λοιπόν λιγότερα πράγματα από όλες μας τις επιτυχίες μας. Εγώ θέλω περισσότερες επιτυχίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Δεν μπορούμε όπως θέλουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε κάθε χρόνο μια νέα κατευθυντήρια γραμμή για την ε, Ευρώπη που τώρα λέγονται Ευρώπη 2020 πριν ήδη ήταν η λεγόμενη στρατηγική της Λισαβόνας να έχουμε όλο και πιο φιλόδοξα έργα από τον ε, αντιδραστήρα σύνδεξη στο ίτερ μέχρι το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Γαλιλαίο. Ταυτόχρονα να λέμε πως δεν θα μεταρρυθμίσουμε τίποτα στη γεωργία, δεν θα αγγίξουμε τίποτα από εκεί πέρα, αλλά θα λάβει λιγότερα λεφτά. Σας λέω από τώρα που θα καταλήξει αυτό το συμπέρασμα σε δραματικές μειώσεις που κάποιοι θέλουν για την πολιτική συνοχής. Οπότε θα, ε, δεν χρειάζεται νομίζω να σας περιγράψω την περαιτέρω απίσχναση και διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα για το 2012 έχουμε συν 10 ε, δισεκατομμύρια ευρώ για έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί και θα εκτελεστούν και έχουν υπογραφεί, τα οποία δεν θα εκταμιευτούν. Και θα εξασληθούν τα κονδύλια τον Σεπτέμβριο ήδη. Συγκεκριμένα, δηλαδή με τις προοπτικές που μας δίνουν ήδη αρχηγοί Καρδών και κυβερνήσεων και ακολουθούν τώρα ως πολιτικοί, μπορώ να σας πω μόνο ένα πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί ήδη να πληρώσει τους λογαριασμούς τους για μέτρα που έχουν ληφθεί σε πολλές περιφέρειες. Γιατί οι απαιτήσει οι διάφορες δεν προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Από τα κράτη-μέλη προέρχονται. Και ποιος αρνείται να δώσει τα λεφτά για να πληρωθούν οι λογαριασμοί για αυτά τα οποία παρήγγειλαν τα κράτη-μέλη, πάλι τα κράτη-μέλη. Ε, δεν μπορεί η δεξιά να αποφασίζει και η αριστερή να αρνείται να πληρώσει. Δεν είναι αυτή η υπεύθυνη πολιτική. Γι' αυτό είναι διατεθειμένο να παλέψει και να διαπραγματευτεί σκληρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ 1993 και 1999, προπολογισμός της Ένωσης κατά μέσο όρο ήταν 1,18% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω το νούμερο. Μεταξύ 1993 και 1999 κατά μέσο όρο, 1,18%. Από το 2000 δε, ο προπολογισμό έπεσε στο 1,06% του ΑΕΠ. Αυτά όσον αφορά την εξοικονόμηση. Είμαστε ένα κοινοβούλιο που κάνει οικονομίες. Και τώρα ζητάνε διάφορες χώρες 1%. Δηλαδή, εάν δούμε και τον πληθωρισμό των τελευταίων ε, ετών, μιλάμε για μία μείωση κατά 15%. Το πιο 15% τώρα των έργων δεν θα υλοποιηθεί, δεν μας το λέει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ένα λοιπόν πρέπει να είναι ξεκάθαρο, κυρίε και κύριοι με μεγάλες περικοπές και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι δυνατόν να κάνουμε μια λογική πολιτική επενδύσεων. Η Ευρώπη όμως χρειάζεται ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και δουλειές. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε στην απέτησή μας για έναν ανάλογο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Κυρίε και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περιφερειές, οι πόλεις είναι συνεταίροι και προσπαθούν να βρουν μια διέξοδο από την κρίση. Όλοι, εμείς και εσείς, εδώ στο Κοινοβούλιο, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλοι υπηρετούμε τους πολίτες της Ευρώπης. Και αυτό μας υποχρεώνει να είμαστε αλληλέγγυοι και παρακολουθώ μεγάλη ανησυχία πως η κρίση αυτή στην οποία βρισκόμαστε κινητοποιεί φυγόκεντρες δυνάμεις στην Ευρώπη που οδηγούν σε κατάργηση της ελεγγύης. Χωρίζεται ή τουλάχιστον κινδυνεύει να χωριστεί η Ευρωπαϊκή μας Ένωση σε βορρά εναντίον νότου, ανατολή εναντίον δύσης, ε, σε πλούσιους εναντίον φτωχών και στο τέλος ένα είναι σαφές. Είτε όλοι μαζί θα κερδίσουμε, είτε όλοι μαζί θα χάσουμε. Γιατί βεβαίω εν τη ενώση η δυνάμει. Εύχομαι σήμερα λοιπόν να έχετε επιτυχείς διαβουλεύσεις και θα ήθελα εδώ πέρα να ευχαριστήσω ρητός για την να σας ευχαριστήσω ρητός για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να μιλήσω στην αρχή των εργασιών σας. Όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Χέρμαν Φαν γιατί βεβαίως διαπιστώνουμε πως δεν είναι ε, ο αρχηγός, ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτός τον οποίο ασκώ κριτική, αλλά οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ο Δε Χέρμαν ότι είναι πολύ καλός συνομιλητής για τα προβλήματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό βεβαίως ισχύει και για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οπωσδήποτε για τους εκπροσώπους της Κυπριακής Προεδρίας που σε αυτή τη δύσκολη φάση καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες. Για την Ντανούτα Χίμπνερ δε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω τίποτα. Και το ότι βεβαίως έχουμε και πρόεδρο τον πρόεδρο μιας ε, ισπανικής περιφέρειας σημαίνει πως πρέπει νομίζω να καταβάλουμε προσπάθειες από κοινού εντός των χωρών μας και μεταξύ των χωρών μας για να βγούμε από την κρίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ήρθατε εδώ και για όλα όσα μας είπατε. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να λάβει το λόγο. Of the European Parliament, Tia Martin, Mr. President of the Committee of the Regions, Mr. Valcarcel, Mr. President of Chair of the European Parliament's Regional Policy Committee, Mrs. Hübner, Madam Minister,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 και, αλλά θα πρέπει παράλληλα να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την αναπτυξιακή αυτή πορεία. Θα πρέπει η Ευρώπη να είναι δελεαστική ήπειρος όπου να μπορεί κανείς να ζει, να εργάζεται και να δημιουργεί πλούτο καθώς και να τον δαπανά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ανάπτυξη, ποιοτική ανάπτυξη και έναν διάλογο περί συνοχής και δικαιοσύνης. Από το 2008 είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύο αλληλένδετες κρίσεις, ε, την τραπεζική κρίση και την κρίση των ε, εθνικών χρεών. Όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν συγκλονιστικές επιπτώσεις, πολύ περισσότερες από αυτές που είδαμε. Και είδαμε ότι δημιούργησαν μεγάλους κλειδονισμούς σε πολλές χώρες. Όλα αυτά όμως είναι ευπρόσδεκτα κατά κάποιο τρόπο, διότι οι δημόσιες αρχές συνδράμουν για να βοηθήσουν τις χώρες που αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες, να ε, δημιουργηθούν ρυθμιστικές αρχές για τις τράπεζες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτούς τους κλειδονισμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντιγνωμίες, ούτε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όμως η Ήπειρός μας θα μπορούσε να οδηγηθεί σε πλήρη καταστροφή. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η δημοσιονομική εξυγίανση δεν είναι στόχος αφεαυτού. Θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να δούμε αυτή τη δυναμική πορεία της αγοράς. Βλέπουμε ότι τα επιτόκια αυξάνονται, η ζήτηση μειώνεται και ανακύπτει η κρίση. Το ζήτημα όμως είναι πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την εξυγίανση που είναι αναπόφευκτη κατά έξυπνο, κατά ευφύ τρόπο, έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι ο βασικός μοχλός αντιμετώπισης και πολλές χώρες έχουν αναλάβει αυτή τη διαδικασία μέσα στα πλαίσια των επενδύσεων και της απασχόλησης. Και ε, μάθαμε ότι αυτοί που το κατάφεραν στο παρελθόν, όπως η Γερμανία 10 χρόνια πριν και η Φινλανδία και η Σουηδία 20 χρόνια πριν, τα κατάφεραν πολύ καλά. Έχουμε πολύ ενθαρρυντικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη έτσι ώστε να προωθήσουμε τον τομέα της ενέργειας, την αγορά εργασίας και πιστεύω ότι η κοινωνική δικαιοσύνη μπορεί να επιτευχθεί όταν έχουμε ίση κατανομή θυσιών. Έτσι μπορούμε να μάθουμε ημέν από τους δε. Όλοι γνωρίζουμε ότι η αποτυχία ή η επιτυχια μίας χώρας μπορεί να αλλάξει την εικόνα για όλες. Όμως, αυτό που έχει σημασία είναι να εργαστούμε από κοινού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε την ενιαία αγορά. Φτάσαμε σε μεγάλα επιτεύγματα, αλλά μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα μέσα στα πλαίσια της αγοράς ενέργειας και της ψηφιακής αγοράς. Τώρα το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ασχολείται με το θέμα της ψηφιακής αγοράς. Μας ενδιαφέρει και το θέμα των δημόσιων αγορών. Επίσης θα έχουμε ένα δεύτερο πακέτο 12 δράσεων για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις μας στο διεθνή χώρο. Θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι πρόσβασης και το διεθνές εμπόριο, οι διεθνείς συναλλαγές είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη. Έχουμε συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες με πολλές χώρες. Δείτε την κινητικότητα και την κατάρτιση. Παρά τη μεγάλη υποαπασχολησιμότητα έχουμε 2 εκατομμύρια θέσεις προς πλήρωση. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα προγράμματα τύπου Εράσμου και να εντάξουμε ειδικέ γραμμές στον κανονικό μας προϋπολογισμό. Ακόμα και αν πρόκειται για το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, μιλάμε για ένα 3 ευρώ μέσα σε μία επταετία, κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει μεγάλη σημασία στον τομέα της μόχλευσης. Επίσης, θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε εκεί που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν. Γι' αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί και το θέμα των δημοσιονομικών προοπτικών, των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών, κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσει, θα απασχολήσει ένα ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γύρω στο Δεκέμβριο με τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά έχουν συζητηθεί σε διάφορα επίπεδα για περισσότερο από ένα Υπάρχουν διχογνωμίες, αλλά μιλάμε για ένα 0,1% του ΑΕΠ. Και πιστεύω ότι οι 27 αρχηγοί κυβερνήσεων θα μπορέσουν να συμβιβαστούν, να βρουν ένα συμβιβασμό για αυτό το ποσοστό. Κάτι το οποίο είναι χαμηλότερο από άλλα επίμαχα ζητήματα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε το Νοέμβριο ως προς τις ε, πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές, διαφορετικά δεν θα υπάρξει ούτε ανάπτυξη ούτε απασχόληση. Πέρα από τον προϋπολογισμό έχουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είναι η μεγαλύτερη τράπεζα πολυμερών σχέσεων διεθνώς. Τη γνωρίζει το ευρύτερο κοινό και Νομίζω ότι γνωρίζετε ότι ασχολείται και με θέματα υποδομής. Μιλάμε για 10 δις έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα δανειοδότησης μέχρι 60 δις που θα πολλαπλασιαστούν και θα φτάσουν στα 180 δις. Ας δούμε τώρα τις περιφέρειες. Είναι σημαντικοί παράγοντες και φορείς γιατί μέσα στα πλαίσια του νομοθετικού έργου δαπανούν 800 ε, δις και έχει μεγάλη σημασία για τις δημόσιες υπηρεσίες, για τις στρατηγικές ανάπτυξης και ούτω καθεξής να εμπλακούν και στη διαδικασία της Ατζέντα 2020 για να χρησιμοποιηθούν σωστά τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Βεβαίως, οι κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα εθνικά ελλείμματα. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εμπλέξουν και τις περιφέρειες σε αυτή τη διαδικασία. Έχει μεγάλη σημασία η δημοσιονομική εξυγίανση κατά φιλικό, ας το πούμε, τρόπο. Φιλικό προς τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να προωθήσουμε την εργασία, την απασχολητισμότητα γενικότερα. Υπάρχουν πολλά περιθώρια και Μιλάμε για μια κοινή προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης, γιατί μιλάμε για πολυσχηδείς ε, και πολλές πτυχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όπως ξέρετε, οι επιλογές είναι δύσκολες και το διακύβευμα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να αλλάξουμε την πορεία μας διαφορετικά. Αυτό, ε, αν δεν καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το διακύβευμα, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε μας. Οι περικοπές θα πρέπει να είναι δίκαιες. Δεν θα πρέπει τις θυσίες να τις υποστεί μία οικονομική ομάδα ή μία γενιά. Χρειάζονται περισσότερες αλλαγές, διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες είναι όμως χρονοβόρες. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες μας ακριβώς τι προσπαθούμε να καταφέρουμε, θα πρέπει να τους πείσουμε με ε, συγκεκριμένα γεγονότα και στοιχεία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε θετική, μια θετική γλώσσα. Υπάρχει μεγάλος αρνητισμός, φόβος και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια γλώσσα ελπίδας, η οποία θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε τις αλλαγές. Το κάναμε στο παρελθόν, θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε και το μέλλον μας κατά τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Uh, Μια και αποσιάζει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, μας είπαν ότι θα απευθύνει λόγο μέσω βίντεο. Δεν ξέρω αν ε, είμαστε έτοιμοι τώρα να τον ακούσουμε. Mesdames et messieurs, chers amis. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, λυπάμαι που δεν βρίσκομαι μαζί σας σήμερα για την δέκατη διοργάνωση των ανοιχτών ημερών. Ήθελα όμως να απευθυνθώ σε σας μέσω αυτής της βιντεοσκόπησης. Οι Open Days αποτελούν ένα μείζον γεγονός της περιφερειακής πολιτικής. Μία αναγκαία πλατφόρμα συζητήσεων για τον ρόλο της ε, πολιτικής συνοχής μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής αντιμετώπισης της κρίσης και για να αντιμετωπίσουμε την ανάπτυξη του αύριο. Σήμερα είμαστε μεταξύ μας επιχειρηματίες, πολιτικοί, ε, επικεφαλής ε, κυβερνήσεων και προσπαθούμε να φτάσουμε σε μια πιο δυνατή και ενωμένη Ευρώπη ως απότοκο της κρίσης. Θα ήθελα να σας ε, τονίσω λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Χέρμαν Βαν Ρομπόι, και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Μάρτιν Σούλτς, μπορούν να συνδράμουν την Επιτροπή μέσα στα πλαίσια αυτής της εταιρική σχέσης που προωθήκε η Επιτροπή με την Επιτροπή Περιφερειών. Θα πρέπει να καταδείξουμε ότι οι διάφοροι φορείς και θεσμικά όργανα της Ένωσης συνεργάζονται για την συνοχή, για την περιφερειακή ε, πολιτική, για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης, γιατί η εμπιστοσύνη είναι στοιχείο κλειδί της ανάπτυξης, αλλά όλα αυτά δεν θεσμοθετούνται. Θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή πολιτικές που να οδηγήσουν σε μία βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα τρίπτυχο Μιλάμε για τις δημοσιονομικές αλλαγές, τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές και τις στόχοθετημένες επενδύσεις. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση. Η οικονομία της Ευρώπης είναι ευάλωτη και γι' αυτό δεν είναι θετικά τα σημάδια που έχουμε. Θα πρέπει να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Ευρώπη. Σε ορισμένες περιφέρειες είναι δραματική η κατάσταση. Βλέπουμε ότι υπάρχει όλο ένα και περισσότερη φτώχεια. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όμως θα ήταν ε, ιδιαίτερα επιζήμιο να γυρίσουμε στις παλαιές μας συνήθειες που ε, μας οδηγούσαν σε ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης μέχρι τούδε. Δηλαδή, ε, αν, δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχουν οι μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα και για την οικονομική πρόοδο. Δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Θα πρέπει να δράσουμε με συνοχή και αποφασιστικότητα, συνδυάζοντας ε, τις μεταρρυθμίσεις και την κοινωνική δικαιοσύνη μέσα στα πλαίσια και της ευθύνης αλλά και της αλληλεγγύης. Διαθέτουμε μία αναπτυξιακή ατζέντα, τη στρατηγική 2020, για να εξυγχρονίσουμε και να διατηρήσουμε την οικονομία μας, η οποία να βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό ε, μοντέλο. Δεν νομίζω ότι το κοινωνικό μοντέλο έχει αποβιώσει. Δεν συμφωνώ καθόλου. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε και να λάβουμε υπόψη μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δικά μας μέσα και μηχανισμούς. Ένα από αυτά τα μέσα είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Θα θέλαμε να συντάξουμε έναν προϋπολογισμό ανάπτυξης και επενδύσεων για την απασχόληση και την καινοτομία. Βλέπουμε ότι η πολιτική της συνοχής καθίσταται ολοένα και σημαντικότερη μέσα στα πλαίσια των ε, δημοσιονομικών διαδικασιών. Και ακριβώς επειδή ορισμένα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, πολλές φορές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να προωθήσουμε επίσης την ανάκαμψη και την οικονομική συνοχή δεν μιλάμε μόνο για, τις, για χώρες που ευεργετούνται, τις χώρες δικαιούχους όπως τις κατονομάζουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς όλα αυτά θα ενταχθούν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, γιατί πρόκειται για αλληλένδετα μέσα. Από την απαρχή της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά κονδύλια και επιστώσεις να χρησιμοποιηθούν στοχοθετημένα. Γι' αυτό έχουμε αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε νέα κράτη-μέλη και μέσα στα πλαίσια ενός συμπληρώματος βοηθείας για τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση, ήδη 14,5 δις ε, ευρώ έχουν ενταχθεί και έχουν δοθεί, χορηγηθεί προς τις χώρες αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε αυτές τις στοχοθετημένες επενδύσεις που να δημιουργούν ανάπτυξη στο μέρο της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας για να υποστηρίξουμε τις ΜΜΕ. Μεταξύ 2009 και 2012 περίπου 20 δις χρησιμοποιήθηκαν και επαναπρογραμματίστηκαν για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις νέες ανάγκες. Τα κράτη έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την ανεργία των νέων. Γι' αυτό διαθέσαμε 10,4 δις ευρώ για να βοηθήσουμε τους νέους που δεν έχουν εξεύρει ακόμα εργασία. Θα συνεχίσουμε αυτή μας τη δυναμική πορεία. Ο προϋπολογισμός είναι το κατεξοχήν μέσον για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αναπτυξιακή ατζέντα της Ευρώπης 2020 και η συνοχή είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να διέπουν την πολιτική μας χρηματοδότησης. Δεν μιλάμε για τη συνοχή που βρίσκεται από τη μία πλευρά και την ανταγωνιστικότητα που βρίσκεται από την άλλη. Πρόκειται για ένα κοινό μέσο για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, αλλά να δώσουμε και μία νέα πνοή στην ανάπτυξη. Η πολιτική σύνοχης μπορεί να βοηθήσει τις περιφέρειές μας, τις πόλεις μας, τις αγροτικές περιοχές. Όλα αυτά θα πρέπει να ε, επανενταχθούν στο στόχο της ανάπτυξης, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες προκλήσεις. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο ανταποκρινόμαστε στον τομέα της απασχόλησης, για παράδειγμα. Μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τον προσεχή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα όλοι να προσδώσουμε στην Ευρώπη τον προϋπολογισμό που της αξίζει. Πρόκειται για την αξιοπιστία μας και ξέρω ακριβώς τι σας ζητώ θα πρέπει να ζητήσουμε από τους επικεφαλείς των περιφερειών να προωθήσουν, να ε, ορθώσουν το ανάστημά τους και να ενισχύσουν τη δική τους φωνή. Αυτό θα πρέπει να γίνει και στις Βρυξέλλες αλλά και στο Στρασβούργο, μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Γιατί αν υπάρχουν ε, λήψεις ή χάσματα τότε θα βρεθούμε στην άκρη αυτής της διαδικασίας. Δεν μιλάμε για μία συγκεντρωτική πρωτεύουσα που είναι οι Βρυξέλλες. Όλα αυτά υπηρετούν τις περιφέρειες. Γι' αυτό θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί υπάρχει πραγματικά προστιθέμενη αξία που απορρέει από τις επενδύσεις στις οποίες θα προβούμε μέσα στα πλαίσια της ε, πολιτικής συνοχής και της περιφερειακής πολιτικής. Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε εσά. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και θα είμαστε σε επαφή έτσι ώστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προωθήσουμε την πολιτική μας συνοχή στην περιφερειακή πολιτική τους πολίτες μας και μια μεγαλύτερη ευημερία για τους συμπολίτες μας γενικότερα. Uh, και τελευταία θα, ζητήσει το θα λάβει το λόγο η Υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου, τη ασκούσε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Μα... έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ θερμά τους ε, οργανωτές αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης που είναι περίτρανη απόδειξη της ε, καταπληκτική συνέργειες που μπορεί να έχουμε όταν διοργανώνουμε τέτοιου είδου ε, εκδηλώσει και είναι ενδιαφέροντος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Κυπριακή Προεδρία έχει αναλάβει τη δέσμευση να εργαστεί προ μια καλύτερη Ευρώπη, μια Ευρώπη που θα είναι πιο κοντά στους πολίτες και θα είναι προσανατολισμένη προς την ανάπτυξη. Θα είναι το σωστό μείγμα αλληλεγγύης, οράματο, ε, αίσθηση του σκοπού, πειθαρχία και προσήλωση στι θεμελιώδει αρχέ και αξίες μα καθώς και ενίσχυσης του της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφική συνοχής, που είναι βαθιά ριζωμένη στην προσέγγιση μας. Όλα αυτά θα καθοδηγήσουν την προσπάθειά μας. Το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο της περίοδου 2014-2020 βρίσκεται στο επίκεντρο του θεματολογίου και του προγράμματος της ε, Κυπριακής Προεδρία. Είναι η ψηστή μα προτεραιότητα ε, θέλουμε να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε συμφωνία μέχρι τα τέλη του 2012 όπως προβλέπει και, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου. Θέλουμε με το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να εξασφαλίσουμε αρκετού πόρους για να διέλθουμε από την οικονομική κρίση και να προβλέψουμε μια υγιή βάση για τη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας χωρίς ταυτόχρονα να παρακολύουμε την ανάπτυξη. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες που μας εξέφρασε πριν από λίγο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι ένα εργαλείο που θα επαναφέρει στην κατεύθυνση της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι μία άμεση συμφωνία για έναν δίκαιο και αποτελεσματικό προϋπολογισμό αποτελεί θεμελιώδη μας στόχο της ε, Κυπριακής Προεδρίας που είναι ένας έντιμος ε, διαμεσολαβητής και θέλει να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ των ε, διεσταμένων ιδεών και να καταλήξει συμφωνία που θα γίνει δεκτή από όλους. Και σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, τους δύσκολους από οικονομική άποψη, καιρούς όπου επικρατεί η ευεβαιότητα, στόχος μας είναι ακριβώς να αντικατοπτήσουμε την πραγματικότητα της κατάστασης. Ε, και στο πλαίσιο αυτό η, η ιδέα των ποιοτικών δαπανών θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να έχουμε προγράμματα με γνήσια θεμενή αξία και αυτά να χρηματοδοτούμε. Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Νοεμβρίου όπως προανέφερε και ο πρόεδρος Βαν Ρομπόι, θα έχει κεφαλαιώδη σημασία μια και θα αφιερωθεί αποκλειστικά και μόνο στην ε, συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η σοβούσα ε, χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μας δίνει ε, τροφή για σκέψη προκειμένου να δούμε πώς θα ε, δώσουμε έμφαση χάρη στην συνεργασία με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση. Και με την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες θα διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η προτινόμενη νέα πολιτική συνοχή στόχο έχει την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ο πρωταρχικός σκοπός της πολιτικής πολιτική συνοχής είναι να μειώσει τις κοινωνικές, οικονομικές και εδαφικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και περιφερειών και που ίσως λόγω της κρίσης ε, εντάθηκαν. Η πολιτική συνοχής είναι η πιο απτή απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και βασικός της στόχος θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι ε, το να φέρει τους Ευρωπαίους πολίτες πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο κοντά μεταξύ τους. Στόχο έχει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε περιφέρειας και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προκειμένου η διαφορετικότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών να αξιοποιηθεί και να μετατραπεί σε πλούτο και πλεονέκτημα. Επίσης ε, θα πρέπει και η πολυμορφία να αποτελέσει τον πλούτον μας. Με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση και με απόλυτη συμπερίληψη της εδαφικής διάστασης ε, όπως προβλέπει και η συνθήκη της Λισαβόνας για την πολιτική συνοχή. Η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί ως ύψητη προτεραιότητα την ε, αποτελεσματική διαχείριση της πολιτικής συνοχής. Και σίγουρα ε, η σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα ήδη απέφερε καρπούς. Την επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αναμένεται να ληφθεί συμφωνία για ορισμένα από τα εκρεμή ζητήματα. Και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου ευελπιστούμε ότι θα επιληθούν όλα τα εναπομείναντα ζητήματα και θα διευθετηθούν όλες οι εκκρεμότητες. Επίσης η Κυπριακή Προεδρία έχει ξεκινήσει τον άτυπο τριμερή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της Προεδρίας είναι να καταλήξει σε μία συνεννόηση και μία κοινή αντίληψη όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων για θέματα προγραμματισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί βεβαιότητα στις περιφέρειες και στα κρατημέλη στην προσπάθειά τους να καταρτήσουν τα νέα τους προγράμματα. Κυρίες και κύριοι, οι περιφέρειες διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μια παραδοσιακή, ε, κλαδική, κεντρική, συγκεντρωτική προσέγγιση πολλές φορές έχει αποτύχει στην αντιμετώπιση των ιδιαζών των προβλημάτων των διαφόρων περιφερειών. Μια νέα πολιτική και νέα διακυβέρνηση προϋποθέτει καλύτερη χρήση του τοπικού δυναμικού ε, για να προσαρμόζει τις επενδύσεις στις τοπικές ανάγκες, να βελτιώσει τις, ε, την παροχή των υπηρεσιών και να κινητοποιήσει και το ιδιωτικό κεφάλαιο. Κάτι που προϋποθέτει ένα νέο ρόλο και για τις τοπικές και για τις περιφερειακές και τις εθνικές αρχές. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ τους και να δοθεί νέα ε, έμφαση στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην επικοδομητική δηλαδή και καρποφόρα ε, αλληλεπίδραση των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών φορέων και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε στην τοπική γνώση, στον τοπικό προγραμματισμό, εφαρμογή και παρακολούθηση προσπαθώντας να εφαρμόσουμε την πολιτική Ευρώπη του 2020 για μια ευφυή, βιώσιμη οικονομία που δεν θα αποκλείει κανέναν. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα μέσα στη, τοπική αυτοδιοίκηση για να εφαρμόσουν τις αντίστοιχες εθνικές στρατηγικές. Και μέσα στα εθνικά πλαίσια θα πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να, που ορισμού γνωρίζει καλύτερα τις τοπικές ανάγκες και τις ε, τοπικές απειλές και τα δικαιώματα, να, να μπορεί και αυτή να υλοποιήσει τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Και στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής μπορεί να ευνοήσει και να προωθήσει περισσότερο τις προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης με μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, προκειμένου να ε, προωθήσει και την οικονομική ανάπτυξη. Ίσως ήρθε η ώρα να, να θεωρήσουμε το πεδίο εφαρμογής ε, και το μέγεθος των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για να δούμε πώς θα πρέπει οι τοπικές στρατηγικές να οργανωθούν και να τύχουν διαχείρισης και αξιολόγησης. Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι οι διάφορες πόλεις και περιφέρειες ε, έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και ως προς το δυναμικό της οικονομικής τους ανάπτυξης, αλλά είναι διαφορετικές και οι προσπάθειες που καταβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προσπαθώντας να απλουστεύσουμε τις κοινοτικέ ε, πολιτικές και την πολιτική συνοχή. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να υπογραμμίσω τον σημαντικό ρόλο της πανευρωπαϊκής συνεργασίας των ευρωπαϊκών περιφερειών των ευρωπαϊκών πόλων και των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών. Σήμερα η πανευρωπαϊκή αυτή συνεργασία αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η συνεργασία, η διαπεριφερειακή συνεργασία θα αποτελέσει ισχυρό εργαλείο και τη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που θα συμβάλλει και στην υλοποίηση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω τη σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία που είναι σημαντικό στόχο τη πολιτική συνοχή. Η Κυπριακή Προεδρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ε, ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει την διαπεριφερειακή αυτή συνεργασία στον, στη νέα περίοδο προγραμματισμού να είναι τέτοιο το νομικό πλαίσιο που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητά της. Συνεργασία λοιπόν και διάλογος μεταξύ μας αλλά και με μεταξύ των πολιτών μας, των συμπολιτών μας. Αυτές είναι λέξεις κλειδιά. Αγαπητοί φίλοι, λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστώ. Τι συνάδελφοι μόλις είπα στον πρόεδρο Φαν Ρόμπαϊ ε, πως ακόμα και αν θέλει να μείνει χρειαζόμαστε τη θέση του στο Προεδρείο. Οπότε ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με το δεύτερο μέρος της ε, συνεδρίασης. Έχουμε τώρα την ε, Τζάκι Ντέιβις η οποία θα προεδρεύσει. Έχει λιγότερο χρόνο από όσο ήθελε. Ελπίζω να τη στάσει. Ευχαριστώ λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Τώρα όπως είπε η κυρία Χίμπνερ περνάμε στο πάνελ με τίτλο «Οικονομική ανάκαμψη, πολιτική συνοχής και στρατηγική της Ευρώπης 2020, ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων». Ακούσαμε ήδη από τις αρχικές παρεμβάσεις πόσο σημαντικό θεωρούν οι ομιλητές μας τον ρόλο των περιφερειών και πόλεων και άρα πόσο σημαντική είναι η πολιτική συνοχής. Σας υπενθυμίζω λοιπόν πως ο τίτλος «Ο Γενικός των Ανοιχτών ημερών» είναι πώς οι πόλεις Ευρώπης και οι περιφερειές θα κάνουν τη διαφορά. Θα συζητήσουμε πώς θα κάνουν τη διαφορά, πόση περισσότερη διαφορά μπορούν να κάνουν, τι στήριξη θέλουν και πολλά από τα ζητήματα που ανέφεραν οι ομιλητές μας. Οι ομιλητές μας λοιπόν είναι, ξεκινάμε από εκεί, δίπλα στην κυρία Χιούμπνερ, από τον Ραμόν Βαρκαθέλ Σίζελ, ε, πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών. Στα αριστερά μου είναι ο Γιωχάνες Χάν, Ευρωπαϊο Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτική και η Ντανούτα Χιούμπνερ βεβαίω, πρόεδρο τη Αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι Τζάκι Ντέιβι και θα φροντίσω να έχουμε μια ζωντανή συζήτηση με χρόνο ελπίζω για σχόλια και ερωτήσεις επίσης. Να σας υπενθυμίσω σε όσους βλέπετε από το διαδίκτυο μπορείτε μέσω Twitter και του hashtag ε, EU Open Days να στείλετε μια ερώτηση και μέσα στην αίθουσα υπάρχουν φύλλα για να γράψετε ερωτήσεις. Ε, παρακαλώ λοιπόν γράψτε σύντομες ερωτήσεις και θα απαντήσουμε. Και στο βάθος εκεί πέρα αν θέλετε ελάτε μπροστά να φτάσετε σε ένα μικρόφωνο. Ας ξεκινήσουμε. Ο καφές σερβίρεται. Δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κάθε μιλητή να μην μιλήσει παραπάνω από 7 λεπτά. Θα τηρήσουμε το χρόνο και να σας ε, εξηγήσουν σύμφωνα με τον τίτλο πώς βλέπουν τον ρόλο των περιφερειών και των πόλων σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας για να έχουμε ανάπτυξη και δουλειέ και το τι σημαίνουν όλα αυτά για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής. Αμέσως λοιπόν κύριε Πρόεδρε μπορείτε να ξεκινήσετε. Σας ευχαριστώ κυρία Συντονίστρια, αξιότιμη κυρία Χίμπνερ, αξιότιμη Επίτροπε Χάν, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Περιφερειών, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα τελευταία δέκα χρόνια, Open Days, η εκδήλωση αυτή έχει αναχθεί σε εβδομάδα αναφοράς στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Για τα κοινοτικά θεσμικά όργανα είναι ένα σημείο κλειδί για να γίνει ένα απολογισμός, να ακούσουμε και να εξακριβώσουμε τις πολιτικές προτάσεις και τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε κατά πόσο προσαρμόζονται αυτές στις πραγματικέ μα ανάγκε. Για τις περιφέρειες και τις ε, πόλεις Ευρώπης, τα, οι Open Days, οι ανοιχτές αυτές οι μέρες, είναι ευκαιρία για να εξακριβώσουμε κατά πόσο κάποιες πολιτικές ε, ε, είναι αποτελεσματικές σε ορισμένες πολιτικές, για να ανταλλαγή των, των, των εμπειριών μας, έχουμε νέες επαφές και δημιουργούμε νέα δίκτυα. Διανύουμε κρίσιμες στιγμές για το μέλλον της Ευρώπης και των περιφερειών τους. Σε λίγες εβδομάδες, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφασίσουν για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις ακούσαμε τις ομιλίες των Προέδρων Σούλτς, Βαν Ρομπόι και της ε, Υπουργού της Κυπριακής Προεδρίας, της κυρίας Μαύρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την παρουσία τους στη σημαντική αυτή εκδήλωση. Η παρουσία των υψηλότερων παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την εβδομάδα των πόλεων και των περιφερειών ένα πράγμα μόνο μπορεί να σημαίνει. Το ότι Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα κέριο εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Περιφερειών, ε, ελπίζουμε οι αποφάσεις των αρχηγών ε, κρατών και κυβερνήσεων τις επόμενες εβδομάδες θα είναι συνεπείς αλλά και σύμφωνες με τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τις ποιοτικέ θέσεις εργασίας. Θα πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας επί των ακόλουθων αρχών. Καταρχήν θα πρέπει να εστιάσουμε τις επενδύσεις μας σε σχέδια και προγράμματα που θα ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τρίτον, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ευνοεί την εδαφική συνοχή και να επιτρέπει στις πόλεις και τις περιφέρειες να εποφελούνται από την εσωτερική αγωνά. Γνωρίζουμε ότι η αποτυχία στην υλοποίηση αυτών αποτελεσμάτων ή ασυνέπεια μερικές φορές ε, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις για το μελλοντικό κοινοτικό προπολογισμό δεν θα γίνουν αντιληπτέ ούτε από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ούτε από του πολιτικού εκπροσώπου. Και σίγουρα μια τέτοια αποτυχία στην υλοποίηση των αποτελεσμάτων δεν θα γίνει που δεν αποδεκτή από του Ευρωπαίου πολίτε. Η Επιτροπή των Περιφερειών ήταν απερίφραστη στον τομέα αυτό. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη και έχουμε ανάγκη από μια Ευρώπη που θα προωθεί και την ευθύνη αλλά ταυτόχρονα και την αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που θα δίνει ελπίδε, που θα φέρνει κοντά τους ανθρώπους και θα επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης ξέρουμε, θέλουμε μια Ευρώπη που θα είναι έτοιμη για το μέλλον, θα είναι ανταγωνιστική και ενωτόμα και θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στον κόσμο της ελεξάρτησης του 21ου αιώνα. Ως εκ τούτου από τις ε, διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποδώσουμε στην πολιτική της συνοχής τον μείζον ρόλο του επενδυτικού εργαλείου, όπως ε, της αξίζει άλλωστε. Θα πρέπει επίσης ε, να βοηθήσουμε τις περιφέρειες να στηρίξουν και την απασχόληση και να δημιουργήσουν ε, ανάπτυξη. Γιατί κυρίες και κύριοι, στην ερώτηση υπάρχει εναλλακτική λύση, η απάντηση είναι κατηγορηματική και αρνητική. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Η υποτίμηση του δυναμικού της οικονομικής, κοινωνικής και αδαφικής ε, συνοχής ουσιαστικά θα συρρυκνώσει τις δυνατότητες των περιφερειών μας για να ξεπεράσουν την κρίση. Αύριο η Επιτροπή των Περιφερειών θα εγκρίνει τη γνωμοδότηση για το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο διατρανώνουμε το αίτημά μας για έναν αξιόπιστο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για έναν προϋπολογισμό που θα ξεπερνάει το 1% του ΕΠ. Ένα προϋπολογισμό που θα στηρίζεται σε νέους ίδιους πόρους, που θα έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και που θα χορηγεί την απαραίτητη ευελιξία για την αλλαγή των προτεραιοτήτων ανάλογα με την μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Η ο περιορισμός, η συρρήκνωση του προπολογισμού της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά 95% είναι επενδυτικό προπολογισμό, θα σημαίνει ε, διακινδύνευση των πρώτων δειγμάτων της ανάπτυξη που ήδη παρατηρούμε σε πολλέ από τις περιφέρειές μας πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι η πολιτική συνοχή όχι μόνο βοήθησε στην αύξηση τη ανταγωνιστικότητα των περιφερειών μα και ιδιαίτερα των περιφερειών τη σύγκληση, αλλά ακόμη και οι πιο ανταγωνιστικέ περιφερειέ τη Ένωση επωφελήθηκαν από την πολιτική συνοχή, γιατί έτσι βελτίωσαν την αριστεία του στη συνεργασία που είχαν με τι υπόλοιπε περιφέρειες. Γνωρίζω ότι δεν υπάρχει εύκολη λύση για τη διέξοδο από την κατάσταση αυτή, αλλά ο, οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να εμπλέκει τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς η ε, επικουρικότητα, η σύνδεση και η αναλογικότητα είναι σημαντικά ε, στοιχεία. Και η νέα συμφωνία για την Ευρώπη που πρότεινε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να σέβεται αυτές τις αρχές. Και θα ήθελα να ε, παραλάβω ότι η πολιτική προτεραιότητα κατά την Προεδρία μου στην Επιτροπή των Περιφερειών θα είναι η Στρατηγική Ευρώπη 2020, χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια με ευφύ τρόπο για καλύτερες δαπάνες. Από την Επιτροπή των Περιφερειών θα προωθήσουμε μια αποτελεσματική χρήση των ιδιωτικών και δημοσίων κονδυλίων αξιοποιώντας ε, τη συμπληρωματικότητα των διαφόρων ε, ευρωπαϊκών ταμείων και των ε, καινοτομιών, καθώς και των εργαλείων που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σας ευχαριστώ θερμά για τη δέκατη αυτή διοργάνωση των ανοιχτών ημερών, γιατί θα μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε λίγο ακόμη περισσότερο στο κοινό μας πρόγραμμα για μια ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ το να καταλήξουμε σε μια σωστή συμφωνία στην Σύνοδο του Νοεμβρίου. Κύριε Επίτροπε, τώρα να ακούσουμε τις δικές σας σκέψεις για τις ε, ευρωπαϊκές περιφέρειες και τις πόλεις και το πώς θα γίνει η διαφορά. Φαντάζομαι θα μας πείτε και εσείς κάποια πράγματα από αυτά τα οποία ακούσαμε. Πράγματι. Κύριε Πρόεδρε, Ντανούτα, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στον Ραμόν Λούις ε, για τα δέκα θύματα που πέθαναν από τις πλημμύρες στη μούρφια την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μεταφέρετε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των ε, δέκα θυμάτων και θα καταβάλουμε κάθε ε, προσπάθεια για να βοηθήσουμε τη Μούρθια. Σε δύσκολη αυτή στιγμή. Να σας καλωσορίσω επίσης όλους στις ανοιχτές ημέρες, στις φετινές. Πράγματι, έχουμε ε, μια εκδήλωση η οποία αναπτύσσεται εδώ και 10 χρόνια με έξυπνο και αηφόρο τρόπο και ελπίζω η Ευρώπη να έχει γενικώ μια τέτοια ανάπτυξη. Βεβαίω, οι φετινέ ανοιχτέ ημέρε έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμά, αναφέρθηκε ήδη πολλές φορές, Είμαστε κοντά στο τέλος των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό και άρα και του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής. Οπότε είναι η τελευταία καλή ευκαιρία για να στείλουμε ένα μήνυμα ισχυρό από την πλευρά των περιφερειών στα κράτη-μέλη και στον Ευρωπαίο νομοθέτη. Και θα ήθελα να πω πως ε, ήταν η στιγμή να γίνει αυτό, να έρθει στις Βρυξέλλες, αλλά και στις πρωτεύουσές σας να αγωνιστείτε για τα συμφέροντά σας στους υπουργού κορμικών, στους πρωθυπουργού. Οπότε για την ώρα, για τις ερχόμενες εβδομάδες, νομίζω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την, την πρόκληση του πώς θα βγει από την κρίση και θα αποκαταστήσει την ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή εξόδου λοιπόν βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Στα υγιή δημόσια οικονομικά διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και σε στοχευμένες επενδύσεις για δουλειές και ανάπτυξη. Με αυτή τη νέα οικονομική διακυβέρνηση λοιπόν η πολιτική συνοχή πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Έχουμε προχωρήσει αρκετά για να αλλάξει η εικόνα και η σημασία της πολιτικής συνοχής. Θυμάμαι πως όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου δεν είχε τον ρόλο τον οποίο άξιζε η πολιτική συνοχή από τους πολιτικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα μετά από τρία χρόνια η πολιτική συνοχή έχει κεντρικό ρόλο σε όλα τα βασικά έγγραφα, τα οικονομικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας από την πρόταση του προϋπολογισμού, τις συστάσεις αναχώρα, μέχρι το πρόσφατο σύμφωνο ανάπτυξης που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο. Και αυτό κυρίε και κύριοι δικαίω, γιατί από κοινού καταφέραμε να έχουμε μια νέα νοοτροπία όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Η προκάτοχό μου, η Ντανούτα Χίμπνερ, το έκανε αυτό με το να καθορίσει και να δεσμεύσει επενδύσεις ειδικά στο πλαίσιο της ατζέντα της Λισαβόνας. Επίσης θυμάμαι πως ε, υπήρχε μια εμπροσοβαρής πληρωμή των διαρθρωτικών ταμείων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Επίσης αυξήσαμε το ποσοστό συγχρηματοδότησης ειδικά για τις χώρες του προγράμματος βοήθειας για να υπάρξει περαιτέρω ρευστότητα και επίσης προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δώσαμε πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ για αηφόρο ανάπτυξη. Στις ε, υπηρεσίες, στην ε, καινοτομία και ανάπτυξη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, στις υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η φόρο, ενέργεια, μεταφορές και υποδομές ηλεκτρονικές, πολιτικές για την αγορά εργασίας και τις ευπαθείς ομάδες και βεβαίως θα υπάρξει και πρόσβαση χρηματοδότηση για πάνω από 56.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς επίσης και καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, παραδείγματο χάρη μέσω της απόκτησης ε, νέων προσόντων. Επίσης έχει υπάρξει σύμφωνα με τα κράτη-μέλη 210.000 θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργήθηκαν το έτος 2011 που προστίθενται στις υπόλοιπες και φτάνουμε άρα σε ένα σύνολο 405.000 θέσεων εργασία οι οποίε δημιούργηκαν βεβαίω. Αυτέ οι προσπάθειε δεν θα ήταν επιτυχεί χωρί τη δική σα συνεισφορά και την ετοιμότητά σα να δράσετε γρήγορα και έξυπνα και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω γι' αυτό. Αλλά βεβαίω η πολιτική μπορεί και πρέπει να αυξήσει την αποτελεσματικότητά τη. Γι' αυτό προτείναμε για τη νέα πολιτική μετά το 2014 να εγγραφούν αυτές οι αρχές της έξυπνης αηφόρου και με κοινωνική πτυχή ε, ε, επενδύσεων μέσω της θεματικής συγκέντρωσης της αρχής της αιρεσιμότητας να υπάρξουν επίσης σημαντικότερες ε, μεταρρυθμίσεις και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα καθώς επίσης και την ενθάρρυνση διασυνοριακών πρωτοβουλειών συγκεκριμένα στην Βαλτική και στην περιοχή του Δούναβη. Είμαι λοιπόν πεπισμένος πως το σύνολο όλων αυτών θα είναι πως η πολιτική συνοχή θα είναι στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όμως το να είναι βεβαίως στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής σημαίνει και περισσότερες ευθύνες και η πολιτική συνοχή οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή εξετάζεται από όλες τις πλευρές. Πρέπει λοιπόν τώρα να έχουμε αποτελέσματα να κάνουμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε. Να δείξουμε πως τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και πως θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να δημιουργήσουμε δουλειές και ανάπτυξη ειδικά για τους νέους. Και επίσης να επιδείξουμε πως μιλάμε σοβαρά όταν μιλάμε για τη μεταρρύθμιση και την θεματική συγκέντρωση, τα αποτελέσματα και την αρχή της αιρεσιμότητας. Πρέπει να δείξουμε πως μέσω της θεματικής συγκέντρωσης φροντίζουμε να υπάρχει το κατάλληλο μείγμα επενδύσεων. Γνωρίζω πως βεβαίω αυτό μπορεί να μην το θέλουν πάντα οι περιφέρειες, αλλά πιστέψτε με, τα παραδείγματα από το παρελθόν εκεί όπου είχαμε πολλές επενδύσεις στις βασικές υποδομές τις οποίες δεν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως λόγω της έλλειψης επενδύσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έρευνα και ανάπτυξη και μέτρα αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας πρέπει να αποφευχθούν. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μετρήσιμους στόχους και ορόσημα για να αξιολογήσουμε την πρόοδο των προγραμμάτων και να έχουμε μια βάση για μια πραγματική πολιτική συζήτηση επί της ουσίας αντί για ε, διαδικασίες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευση που έχουν ένα σημαντικό ρόλο συγκεκριμένη ανάλυση και συλλογή των σχετικών δεδομένων. Ταυτόχρονα πρέπει να τονίσουμε τη συνεισφορά μας στην ανάπτυξη και τις δουλειές μέσω του συστήματος της αίρεσιμότητας καθώς και την πρότασή μας για τη μεταρρύθμιση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ξέρω πως κάποιοι έχετε επιφυλάξει όσον αφορά κάποιες πτυχές αυτών των αρχών, αλλά θα ήθελα να σας πω πως αυτές οι αρχές είναι ο πυρήνα μεταρρύθμισης και αντικατοπτρίζουν το βασικό ερώτημα. Να ζει κανείς ή να μην ζει. Εάν λοιπόν δεν είμαστε αξιόπιστοι σε όλα αυτά, διατρέχουμε τον κίνδυνο η πολιτική να χάσει την σημασία της, κάτι το οποίο κανείς δεν θέλει και βεβαίω καμία περιφέρεια ή κράτος μέλος δεν έχει πραγματικά την πολυτέλεια να το κάνει. Η πολιτική της συνοχής σε κάποια κράτη-μέλη είναι πάνω από το 50% των δημοσίων επενδύσεων και εγγυημένε μάλιστα για μια περίοδο 7 ετών. Δεν ξέρω, κάποιον εθνικό ή περιφερειακό προπολογισμό που έχει τόσο μεγάλο βάθος χρόνου. Και πιο σημαντικό, υπάρχει μια εγγύηση η οποία προσελκύει και περαιτέρω ιδιωτικέ επενδύσεις. Η θεματική λοιπόν συγκέντρωση, η αιρεσιμότητα και τα αποτελέσματα με βάση μετρήσιμους στόχους και ορόσημα είναι αυτά τα οποία θα μας βοηθήσουν για να προωθήσουμε αυτή τη σημαντική πολιτική. Σε λίγα χρόνια η νέα συζήτηση για τον προπολογισμό θα ξεκινήσει. Πρέπει να σκεφτόμαστε ήδη πέρα από το 2020. Γι' αυτό ήταν τόσο σημαντικό για εμένα να εδρεώσουμε αυτή την πολιτική. Ο ρόλος και οι στόχοι της πολιτικής συνοχής αλλάζουν. Πολιτική συνοχής δεν βοηθάει μόνο τις φτωχότερες περιφέρειες, έχει επιπλέον το επιπρόσθετο καθήκον να εφαρμόσει τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης πανευρωπαϊκά, δίνοντας κίνητρα σε όλες τις περιφέρειες. Η αρχιτεκτονική αυτή λοιπόν λαμβάνει υπόψη αυτό το σκεπτικό με το να ενσωματώνει όλε τι περιφέρειες, ανεπτυγμένες, λιγότερο ανεπτυγμένε και αυτές που είναι σε μετάβαση. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως δεν θα βοηθήσουμε περισσότερο τις φτωχέ περιφέρειες. Υπενθυμίζω εδώ πέρα πω 70% του προπολογισμού πηγαίνει στις φτωχέ περιφέρειες. Οι φτωχέ αυτές τι περιφέρειες είναι ευτυχώ, μόνο 25% των περιφερειών και γύρω στο 25% επίσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού των Ευρωπαίων πολιτών. Αλλά κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό είναι να αντιληφθούμε πως καμία περιφέρεια δεν έχει εγγύηση ευημερία. Σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει γρήγορα, οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη εκτίθενται γρήγορα σε νέες προκλήσεις. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά πως η Φιλανδία είχε πολύ σοβαρή οικονομική κρίση ε, το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990, κυρίως λόγω της κατάρρευσης του εμπορίου με την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μέσα σε τέσσερα χρόνια είχε μειωθεί ε, περισσότερο από 10% η παραγωγή και είχε τετραπλασιαστεί το ποστό ενεργείας, έφτασε στο 17%. Η Φιλανδία εφάρμοσε δραστικά μέτρα για τα δημόσια οικονομικά, αλλά αυξήθηκαν οι δαπάνε για έρευνα και ανάπτυξη αποφάσισε η κυβέρνηση να επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση. Και άρα υπήρχαν κίνητρα για διαρθρωτικές αλλαγέ, αυξήθηκε η ανταγωνιστικότητα και η φιλανδική οικονομία μπήκε σε ένα δρόμο ισχυρότερης ανάπτυξης με βάση τη γνώση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περαιτέρω επενδύσει σε αυτόν τον τομέα. Αυτά τα είπαν οι συνάδελφοι. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουν, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις εβδομάδες που έχουμε και ο πρόεδρος του που ήταν σαφής γιατί έχουμε και το έκτακτο συμβούλιο τον Νοέμβριο και πρέπει να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που μένει μπροστά μας και ελπίζω αυτές οι ανοιχτές ημέρες να οδηγήσουν όπως είπα στην αρχή της παρέμβασής μου σε μια εκδήλωση η οποία θα στείλει το μήνυμα των πόλων και των περιφερειών στην Ευρώπη ότι χρειαζόμαστε αυτόν τον προπολογισμό επενδύσεων για να στείλουμε ένα μήνυμα και στους λαούς και στις αγορές για να ξεκινήσουν και οι απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις για να υπάρξουν δουλειές και ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε, πολλά έχουμε να συζητήσουμε, αλλά έπρεπε εσείς να δώσετε το εναρκτήριο λάκτισμα. Και αυτό ακριβώς μας απασχολεί, δηλαδή να δούμε το θέμα του προϋπολογισμού για να πείσουμε και το σύμβουλο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χούμπνερ για να μας μιλήσει για τις δικές της σκέψεις. Πολλά ελέγχθησαν, ε, λέει η κυρία Χούμπνερ, αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσει η μελλοντική πολιτική συνοχή μέσα στα πλαίσια αυτών των ε, κατευθυντηρίων γραμμών. Δηλαδή να έχουμε καλά χρηστά δημόσια οικονομικά, ε, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν κατάλληλες επενδύσεις στην απασχολησιμότητα και να δούμε τι θα γίνει και με τον, ε, με τους, ε, με τον προϋπολογισμό μας μέσα στα πλαίσια βεβαίως των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα γίνουν σε επίπεδο κρατών μελών και να δούμε και την εξάντε αιρεσιμότητα που διέπει αυτό το σχήμα έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη, περισσότερη δράση. Επίσης, θα πρέπει να πούμε, θα πρέπει να τονίσουμε, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης για την αναπτυξιακή αυτή πορεία και θα πρέπει να δράσουμε από κοινού γιατί που οδηγούν στην ανάπτυξη δεν δημιουργούν και τους κατάλληλους όρους προς αυτήν. Χρειάζεται μία γενικότερη σύνδρομη για να φτάσουμε στην σύγκληση αυτή που είναι προαπαιτούμενο για να αντιμετωπίσουμε και την ε, αλληλεξάρτητη αυτή πορεία μας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι η πολιτική συνοχής είναι μία πολιτική επενδύσεων, αλλά θα ήθελα επιπλέον να πω ότι η πολιτική συνοχής 14-20 έχει μεγάλη σημασία ως προς το πώς διαρθρώνεται πώς θα τη διαχειριστούμε, πώς θα έχουμε μία πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και στοχοθετημένες δράσεις. Εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο επενδύσεων για την περίοδο 14-20. Αυτό σημαίνει ότι θα διαπραγματευτούμε το πολιετές αυτό πλαίσιο και θα πρέπει να συνδράμει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο αυτό πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίσει πολλά χρηματοοικονομικά κίνητρα και κίνητρα για αλλαγές. Έχουμε να κάνουμε με μία πολιτική εμπροστοφυλακής Αρχικά είχε οριστεί το 2005-2006, αλλά θα πρέπει όταν συζητούμε για τους στρατηγικούς στόχους 14-20 να κοιτάξουμε και πέραν από το 20, γιατί αυτό έχει σημασία μέσα στα πλαίσια της επιχειρησιακή μας, επιχειρησιακής μας πορείας. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εντάξουμε αυτή τη στρατηγική σε περιφερειακούς και τοπικούς στόχους, έτσι ώστε να υπάρχει ένα αναπτυξιακό πλαίσιο για τις ε, περιφέρειες. Πρόκειται για μια δημόσια πολιτική που θα είναι καταλήτης και υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Άρα υπάρχει δυνατότητα μόχλευσης και αποτελεί και ένα μεγάλο δέλεαρ για τον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να ενταχθεί στο ρυθμιστικό μας πλαίσιο έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος, ο επενδυτικός κίνδυνος. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους όρους για τη συνδρομή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εάν τα διαρθρωτικά ταμεία προωθήσουν αυτές τις αλλαγές μέσα στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και εάν λάβουμε υπόψη τις εδαφικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, θα πρέπει να υπάρχουν ευφυείς περιφερειακές στρατηγικές έτσι ώστε να συνδυαστούν αυτές οι δράσεις. Εάν θέλουμε να λάβουμε υπόψη σοβαρά την εδαφική ιδιαιτερότητα, θα πρέπει να εντάξουμε αυτή την πολιτική σε μια γενικότερη πολιτική συγχρηματοδότησης Διαφορετικά δεν θα ανταποκριθούμε ως προς τις ε, ιδιαιτερότητες αυτές. Ως προς τις επενδύσεις θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει οι πολιτικοί να μπορέσουν να υποστηρίξουν παράγοντες ανάπτυξης που ενέχουν κινδύνους Εάν δεν εντάξουμε και αυτόν τον υψηλό κίνδυνο ως προς επενδύσεις, τότε δεν θα λάβουμε υπόψη σωστά τις ε, προτεραιότητές μας. Αυτή η επενδυτική πολιτική έχει νόημα όταν υπάρχει πρόσβαση στις επενδύσεις μέσα στα πλαίσια ενός πλήρους κύκλου και στα πλαίσια της αιρεσιμότητας. Εάν λοιπόν το, τα κονδύλια συνοχής θέλουμε να τα επεκτείνουμε σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να ενισχύσουμε έναν πλήρη επενδυτικό κύκλο. Θα πρέπει να εντάξουμε αυτούς τους στόχους. Όταν μιλάμε για συμβασμούς, Τζάκι, λυπάμαι, πρέπει να πω δύο πράγματα ακόμα. Υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Αυτή η διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης δυστυχώς οδηγεί σε συρρήκνωση επενδύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό είναι μεγάλο πρόσκομα για το μέλλον. Πολλοί πιστεύουν ότι ό,τι είναι συγκεντρωτικό ενέχει χαμηλότερο κόστος. Θεωρώ όμως ότι η αποκέντρωση είναι σημαντική. Επίσης, ε, στα πλαίσια των προοπτικών 14-20 θα πρέπει να δούμε τον επίγοντα χαρακτήρα αυτού του σχήματος. Τον Οκτώβριο θα προωθηθεί αυτή η διαδικασία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τον Νοέμβριο. Είναι μεγάλη η πρόκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Γνωρίζουμε όλοι τη δυσχέρεια της κατάστασης. Πολλοί ζήτησαν το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε καθυστερήσει, γι' αυτό θα ήθελα να είσαστε πολύ πειθαρχημένοι. Πριν προχωρήσουμε, ο Μάρτιν Σούλς στις αρχικές του δηλώσεις μίλησε για τους φίλους της πολιτικής συνοχής. Μιλάμε για αυτούς τους φίλους ε, της, της συνοχής έναντι αυτών που πιστεύουν στις, σε μια γενικότερη πολιτική δαπανών. Επίτροποι Επίτροπε, ίσως θα μπορούσατε εσείς να μας απαντήσετε. Το καλό μήνυμα λοιπόν είναι πως υπάρχουν μόνο φίλοι εδώ πέρα και κανένας εχθρός. Και νομίζω πως μπορεί να γίνει μια συγχώνευση των δύο αυτών ομάδων ε, φίλων και θα είναι οι φίλοι της ε, ανάπτυξης. Και νομίζω πως αυτό είναι το καλό μήνυμα. Ε, για να σοβαρευτούμε, δεν υπάρχει κάποια αντίφαση. Το ένα σημαίνει έξυπνες επενδύσεις και το άλλο σημαίνει οι έξυπνες επενδύσεις να είναι και αηφόρες και να έχουν αποτελεσματικότητα κτλ. Οπότε δεν υπάρχει κάποια αντίφαση στην πραγματικότητα και νομίζω πως ξεκαθάρισε πως μιλάμε για ένα 0,1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και θα πρέπει νομίζω να στείλουμε τα σωστά μηνύματα στην κατεύθυνση του προπολογισμού που πρότεινε η Κομισιόν, ο οποίος πρέπει να ιδιοθετηθεί τον Νοέμβριο. Σας ευχαριστώ. Οπότε πρέπει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί ε, έτσι το παρουσιάζουν ως το ένα εναντίον του άλλου και εσείς φαντάζομαι θα συμφωνείτε πως δεν είναι σωστή αυτή η ερμηνεία. Εγώ εκπροσωπώ ένα θεσμικό όργανο που πιστεύει, όπως και εγώ πιστεύω ακράδαντα, ότι οι περισσότεροι είναι φίλοι της συνοχής. Εχθροί, αν υπάρχουν, είναι ελάχιστοι, για να μην πω κανένας. Εμείς στην Επιτροπή Περιφερειών ξέρουμε ότι όλες ε, οι περιφέρειες λαμβάνουν κονδύλια. Το θέμα είναι ποιες ε, έχουν ανάγκη για περισσότερα κονδύλια. Πάντως, στην Επιτροπή των Περιφερειών γνωρίζουμε ότι η πολιτική της συνοχής είναι ο ιδεώδης μηχανισμός για να γεφυρώσουμε κάποια κενά και να καλύψουμε τις διαφορές και τις ανισορροπίες που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών. Και δεν είχαμε την Επιτροπή Συνοχής, είχαμε ακόμη πιο πλούσιες και ακόμη πιο φτωχές περιοχές. Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιστορία της ισότητας. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε αυτό το βασικό χαρακτηριστικό. Κύριε Χιούμπνερ, ο Επίτροπο είπε προηγουμένω για την αλλαγή τη νοοτροπία και είπε ότι εσεί πρωτοστατήσατε σε αυτή την αλλαγή τη νοοτροπία. Μήπω όμω τώρα κινδυνεύουμε την κρίση να επανέλθουμε στην παλιά αντίληψη περί πολιτική συνοχή. Μήπω λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώ θα μπορούσαμε να τρέψουμε αυτή την επαναφορά προ το παρελθόν. Ναι, αυτή η συζήτηση είναι πολύ συχνή και τέτοια επιχειρήματα τα ακούμε και στι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό συμφωνώ με τα επιχειρήματα του στρατοπέδου των καλύτερων δαπανών και σίγουρα εδώ και μια δεκαετία ασχολούμαστε με μεταρρυθμίσεις της πολιτικής που στόχο έχουν την πιο αποτελεσματική και την καλύτερη χρήση των κονδυλίων, τον better spending δηλαδή, τον καλύτερο τρόπο χρήσης και αξιοποίηση των δαπανών. Θα πρέπει όμως ε, να συνεχίσουμε αυτόν τον πανευρωπαϊκό διάλογο και να δούμε αν θέλουμε τέτοιες ε, περιφέρειες μετάβασης ή αν θέλουμε αυτό το αποθεματικό των επιδόσεων. Γιατί πιστεύω ότι οι φίλοι της πολιτικής ε, συνοχής είναι αυτοί που πάνω απ' όλα θέλουν την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων. Αυτοί περισσότερο από όλους θέλουν το better spending. Θα πρέπει πάντως να είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση γιατί όπως ξέρετε η πολιτική συνοχή είναι από τις πλέον ε, μεταρρυθμισμένες ή τις πιο συχνά αναθεωρημένες πολιτικές. Και ελπίζω ότι σε κάθε νέα μεταρρυθμίση θα έχουμε και μια καλύτερη ε, πολιτική συνοχής. Ευχαριστώ. Έχω πολλές ερωτήσεις και απορίες, αλλά ζήτησε, το λόγο και συμμετέχοντες ε, στο ακροατήριο. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω και ερωτήσεις από την αίθουσα και από το Twitter. Πρώτα όμως θα δώσω το λόγο στην κυρία Βρέσο, την προηγούμενη πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών και τώρα πρώτη αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, Τζάκη, θα ήθελα εκ μέρους όλων των πολιτικών ομάδων της Επιτροπής των Περιφερειών να μεταφέρω στον πρόεδρο Βαλκάρσελ Σίσο τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, όχι προς τον ίδιο μόνο προσωπικά, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους ε, των περιοχών ε, της Μουρσία, της Ανταλουσίας και της Βαλένσια για τις ε, τρομερές πλημμύρες και το, που προσθέθηκαν στον προηγούμενο τραγικό γεγονός του σεισμού στη Μούρση ιδιαίτερα. Νομίζω ότι χάρη ελεγγύης θα πρέπει να εγκρίνουμε πολιτικές που θα ενισχύουν την ασφάλεια στα ευρωπαϊκά εδάφη και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση και προς αυτή θα πρέπει να ενισχύσουμε και το ρυθμό μας, να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό ε, θα μας ε, βοηθούσε ένας ε, καλός και αποτελεσματικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Είμαι η συγγήτρια της γνωμοδότηση τη Επιτροπής των Περιφερειών για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μάλιστα της αναθεωρημένης γνωμοδότησης ε, που έγινε μετά τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρθηκε ότι φυσικά μας ενδιαφέρει μια καλή συμφωνία. Η οποία να είναι ικανοποιητική για εμάς, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει η συμφωνία αυτή να ισχύει για όλες τις περιφέρειες. Γι' αυτό τασόμαστε υπέρ ενός προϋπολογισμού που μας επιτρέπει να προωθήσουμε την περιφερειακή πολιτική. Λαμβάνοντας υπόψη κάθε τύπο περιφέρειας και να δούμε και θέματα ανταγωνιστικότητας μέσα στα πλαίσια αυτού του μεταβατικού πλαισίου. Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε λοιπόν τα οικονομικά πλαίσια λειτουργίας. Με βάση την έκθεση αυτή που θα ψηφίσουμε αύριο θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το συνολικό ποσό, τα συνολικά ποσά ίσως αποτελούν ένα επενδυτικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορούν να βασιστούν πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες. Εντάχει σας παρακαλώ. Η αρχή της συναπόφασης λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσει, διότι μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο έχουμε να κάνουμε με θέματα που μας αφορούν και δεν έγιναν σωστές διαβουλεύσεις. Επίσης κυκλοφορούν έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν μοιάζουν με το better spending. Δεν υπάρχει καλή, ε, σωστή αποτελεσματικότητα των καλύτερων μορφών δαπάνης. Θα πρέπει να υπάρξει περιφερειακή ολοκλήρωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, αλλά πολλοί θέλουν το λόγο. Βανίστε Ρόι. Ναι, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, καλό θα ήταν να πούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Η Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων είχε λάβει μία έντολη με 4.000 τροπολογίες τότε για να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο. Και αυτό το οποίο θέλουμε βήμα-βήμα είναι να δούμε ολόκληρη την αρχιτεκτονική την οποία υπάρχει και να τη διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Και είναι ξεκάθαρο, αρχές του 2013 πρέπει να έχουμε τις εθνικές εταιρικές συμφωνίες, ετοιμάζονται ήδη οι συμβάσεις από πόλεις και περιφέρειες και βεβαίως εάν δεν ε, έχουμε ολοκληρώσει θα μιλάμε τότε για σέντς και ευρώ και όχι για μέσα. Κατόπιν, οι φίλοι που έχετε εδώ πέρα στο κοινοβούλιο και οι φίλοι των καλύτερων ε, δαπανών και οι φίλοι της συνοχής θα πρέπει νομίζω να συναντηθούν και αυτό θα γίνει παραδείγματο χάρη μέσω της ε, κλίμακας αυτής και της πορείας προς την, ε, την αριστεία. Και αυτό βεβαίως θα γίνει με το να δούμε εξυπνότερα την μετάβαση αυτή το τι απαιτείται για αυτή τη διαδικασία. Και αυτή η συνεισφορά νομίζω πως είναι ουσιαστική και θα έχουμε έτσι καλύτερα ε, επιχειρήματα για να λάβουμε βεβαίω και τα χρήματα τα οποία ζητάμε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω η επόμενη να είναι ακόμη συντομότερη γιατί έχω 25 άτομα εδώ πέρα που θέλουν να μιλήσουν και έχουμε 20 λεπτά και πρέπει να αντιδράσουν και οι ομιλητές μας. Οπότε παρακαλώ όσο δυνατόν πιο σύντομα. Μάικλ Σνάιντερ παρακαλώ. Ε, με συγχωρείτε κάποια τεχνικά προβλήματα. Κύριε Χίμπνερ, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, συζητήσαν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία την Τετάρτη θα συζητήσουμε στην κοινή συνεδρίαση ΚΟΤΕΡ και Επιτροπής ε, Περιφερειών. Τώρα, για το θέμα εδώ πέρα θα ήθελα να πω το εξή συνοψίζοντας. Αυτό το οποίο σκεφτόμαστε εμείς στην ομάδα του ΕΛΚ, αλλά πιθανώς και οι υπόλοιπες ομάδες στην Επιτροπή των Περιφερειών. Χρειαζόμαστε στο μεσοπρόθεσμο αυτό χρηματοδοτικό πλαίσιο αποτελέσματα μέχρι το τέλος του έτους. Είμαστε στις περιφέρειες, στους δήμους πρέπει να προχωρήσουμε τα προγράμματά μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι από πρώτου. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Χρειάζονται λοιπόν γρήγορε αποφάσεις. Οι περιφέρειες θέλουν να συνεισφέρουν για τη στρατηγική του 2020, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα ε, διαρθρωτικά ταμεία για να δημιουργήσουν ανάπτυξη θέση εργασίας. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο εάν πρώτον έχουμε επαρκή κονδύλια αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τον Νοέμβριο και μας ενθάρρυνε νομίζω ο κύριος Φανρόμπο και δεύτερον εάν οι κανόνες για την χρήση ε, των διαρθρωτικών ταμείων μας αφήνουν κάποιο περιθώριο για τις ε, συνολικές αυτές ε, ιδέες όπως είπαμε για την περιφερειακή ανάπτυξη και βέβαια σε αυτό το κενό μεταξύ του 2013 και 2014 πρέπει να αποφευχθεί. Σας ευχαριστώ για Ολμπριχτή. <clears throat> Yes, thank We have here... Εδώ έχουμε ασχοληθεί με τις περιφέρειες και με τις πόλεις. Άρα ή θα είμαστε διπλωματικοί ή θα είμαστε τοπικοί ανοιχτή. Άρα, αφόσον ε, διοργανώσαμε ανοιχτές ημέρες, ας είμαστε ανοιχτοί. Α μην είμαστε και τόσο διπλωματικοί όταν μιλάμε για πολιτική συνοχή. Θα ήθελα να πω ότι από πλευράς βουλευτών υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των φίλων της συνοχής και των φίλων του better spending. Ε, δεν ε, είναι ευτυχής ο ορισμός, διότι όπως είπε και η πρόεδρος μας, η Ντανούτα Χούμπνερ, η μία ομάδα θέλει περισσότερα χρήματα για την πολιτική συνοχής και η άλλη θέλει μείωση των κονδυλίων. Μιλάμε για όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις. Ρωτήστε, ρωτήστε τις ε, κυβερνήσεις σας. Είναι φίλοι της συνοχής ή φίλοι του καλύτερου τρόπου δαπανών, του better spending. Λυπάμαι που δεν ήμουν διπλωματικός, αλλά αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή. Ε, θα πρέπει να είμαστε φίλοι συνοχής, αν θέλουμε ε, συνοχή πραγματικά. Ναι, ευχαριστώ ως συνεισηγήτρια για το Γενικό Κανονισμό. Θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, οι προτάσεις της Κομισιόν ήταν καλές. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο τις βελτίωσε, τις ενίσχυσε δόμικα διαρθρωτικά και θα ήθελα τώρα μαζί με την Κομισιόν να πω στους λεγόμενους ε, φίλους ε, των καλύτερων δαπανών να διαβάσουν την πρόταση. Αν την είχαν διαβάσει και καταλάβει θα ήξεραν πως μπορούν να είναι φίλοι και της συνοχής. Γιατί αυτά τα οποία αναφέρονται εκεί πέρα είναι καλύτερες δαπάνες και αν πραγματικά θέλουμε να βγούμε από την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε αυτά τα επενδυτικά μέσα οι περιφέρειες, ή πόλεις, ή δήμοι. Και δεν φτάνει κάποια οποιαδήποτε απόφαση τον Νοέμβριο. Χρειαζόμαστε μια απόφαση η οποία θα μας δίνει επαρκή μέσα για να κάνουμε πολιτική συνοχή. Οπότε, ως Κοινοβούλιο, εμείς δεν θέλουμε να αποφασίσουμε γρήγορα, θέλουμε να αποφασίσουμε σωστά. Και γι' αυτό, και αυτή είναι η έκκλησή μου εδώ πέρα σε όσους ήρθαν σήμερα από τις περιφέρειες, χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια, το δικό σας lobbying για να έχουμε και τον αναγκαίο προπολογισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λουκ Φαντενμπράντε. Σύντομα παρακαλώ για να ξανακούσουμε το πάνελ και να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ. Δεν είναι συζήτηση μεταξύ καλών και κακών. Για καλή ή κακή πολιτική και καλή πολιτική να είναι ε, αυτό το οποίο θεωρούν κάποιοι. Γιατί βεβαίως εδώ πέρα έχουμε μόνο λόγια, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, συνεταιρισμοί και οι διάφορες συμβάσεις που έχουμε υπογράψει. Αυτά πρέπει να έχουν κάποια ουσία. Και βεβαίως θα πρέπει πέρα από την Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων να δούμε και θέλω να το πω εδώ πέρα όμα πως η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων έχει τελείως διαφορετική αντίληψη και μιλάει για επίπεδα ευθύνη. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθεσεών αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια συνοχή και η έκθεση η οποία προετοιμάζεται για το multi-tier governance να συμφωνεί με η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δηλαδή και με τις δύο διατυπώσεις να συμφωνούν. Επίσης θα πρέπει τα έγγραφα θέσεων να πάνε στα κράτη-μέλη. Και μετά πρέπει η Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού να πείσουμε το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σε λίγο θα σας δώσω το λόγο πάλι στην αίθουσα. Πολλοί υπογράμμισαν αυτά που μας είπαν οι ομιλητές μας από το πάνελ. Αλλά θα ήθελα να δώσετε έμφαση στην ε, ερώτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να δίνετε διακριτική ευχέρεια στις ε, περιφέρειες να λαμβάνουν μέτρα που προσαρμόζονται στις δικές τους ανάγκες πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που θα ανταποκρίνεται στι πολυσχηδεί προκλήσει. Το ακούσαμε και από τον κύριο Σούλτ και από τον πρόεδρο Βαν Ρόμποϊ. Και το θέμα τη ευελιξία βρέθηκε στην στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, όχι για τα οικονομικά, περισσότερο για τι μεταρρυθμίσει. Φαίνεται, ε, κύριε Πρόεδρε, ότι, ε, κύριε Επιτρόπη, ότι είπατε ότι αυτό σχετίζεται με την αξιοπιστία. Ότι αν κάποιο θέλει να κρατήσει τα κονδύλια, θα πρέπει να κρατήσει και τη θεματική συγκέντρωση. Μπορείτε να μας αναπτύξετε αυτή τη σκέψη. Σύντομα, να αφαιρθώ σε κάποια πράγματα τα οποία ακούστηκαν στην συζήτηση. Η θεματική συγκέντρωση δεν είναι ε, αντίφαση με οτιδήποτε άλλο. Έχουμε, αν θέλετε, ε, ένα μενού από το οποίο επιλέγουμε και εμείς λέμε το μενού να αποτελείται από τρία πιάτα και όχι από οχτώ πιάτα. Να έχουμε μία δίαιτα, αν θέλετε, αλλά να μην είναι υπερβολική. Αυτή είναι η λογική της θεματικής επικέντρωσης. Να συγκεντρωθούμε σε κάποια πράγματα, λίγα και καλά. Αλλά το δεύτερο και είναι σημαντικό, εγώ δεν βλέπω κάποια αντίφαση και αντίθεση μεταξύ των δύο ε, επιτροπών ε, του Κοινοβουλίου αλλά και της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω και τις δύο να τις ευχαριστήσω για το ότι έλαβαν υπόψη τις προτάσεις μας. Είναι παντού μπροστά, μπροστά η πολιτική ε, των περιφερειών. Δεν θέλω να ασκήσω κριτική στη, σε αυτούς που ασχολούνται με τη γεωργική πολιτική αλλά εμείς είχαμε δώσει την έκθεσή μας πριν από το καλοκαίρι. Οπότε εμείς κάνουμε τις προτάσεις μας και τώρα αναμένουμε τις οικονομικές αποφάσεις. Και αυτό το οποίο επίσης θέλω να επισημάνω και απευθύνω έκκληση σε όλες τις περιφέρειες. Μην υπάρχει διέρη και βασίλευε. Γιατί κάποιοι σκέφτονται πως αν υπάρχουν περισσότερες ε, περιοχές ε, και περισσότερες περικοπές, θα γίνουν περισσότερες περικοπές στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Εάν δηλαδή έχουμε ένα 25% ε, των περιφερειών που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες και λαμβάνουν πάνω από 70% κονδυλίων νομίζω είναι δίκαιο. Έτσι αντιλαμβανόμαστε την πολιτική. Αλλά βεβαίω αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι και σας παρακαλώ τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να ε, τηρήσουμε αυτή τη γραμμή. Ευχαριστώ. Ε, με κίνδυνο να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Συμφωνώ με αυτά που μας είπε ο κύριος Χάν, γιατί είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και προηγουμένως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικώ θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσαμε το, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω του Πρόεδρου του κ. Σούλτς και ακούσαμε και εκπροσώπους περιφερειών. Όλοι συμφωνούμε ότι η πολιτική συνοχή έχει πολύ περισσότερους φίλους από ό,τι εχθρούς. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να ανοίγουμε χάσματα, ούτε θα πρέπει να δημιουργούμε αντιπαλότητα. Γιατί ποιος θα μπορούσε να είναι κατά της έξυπνης δαπάνης και των χρήσιμων δαπανών. Ποιος είναι δυνατόν να είναι κατά τον, α, της σωστής αξιοποίησης και των έξυπνων δαπανών. Όλοι είμαστε υπέρ των έξυπνων δαπανών και όλοι είμαστε υπέρ της συνοχής. Δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί να γίνομαι αντιπαθητικός. Αυτό που με ανησυχεί όμως με το θέμα των έξυπνων δαπανών είναι ότι σαν να δημιουργούμε μακροοικονομική ρεσιμότητα. γιατί τουλάχιστον με αυτό μοιάζει. Και εδώ θα ήθελα να σταματήσω και να δώσω κάποια τροφή για συζήτηση περαιτέρω. Κύριε Χιούμπνερ, ναι, το θέμα της θεματικής συγκέντρωσης. Γενικώ γίνονται πολλές συζητήσεις στην Επιτροπή και με την Επιτροπή. Δεν είναι πρώτη φορά που ακούγεται αυτό το θέμα. Σας διαβεβαιώ ότι γίνονται εκτενείς συζητήσεις. Και σίγουρα έχουμε τεράστια ανάγκη εξυγχρονισμού, αλλά δεν έχουμε αρκετά κονδύλια στην Ευρώπη. Οπότε η συγκέντρωση είναι επιτακτική ανάγκη. Το θέμα δεν είναι μόνο να προσδιορίσουμε τους στόχους της πολιτικής του 2020 και να την να προσαρμόσουμε στις διάφορες πολιτικές. Θέλουμε απλώς ε, να την προσαρμόσουμε στις ε, διάφορες ανάγκες και τις καταστάσεις, ε, γιατί έχουμε λίγα κονδύλια στον κοινοτικό προϋπολογισμό, οπότε χρειαζόμαστε τη συγκέντρωση. Αλλά θα πρέπει η συγκέντρωση, η επικέντρωση να γίνει στις στοιχειώδεις ανάγκες των περιφερειών. Θα πρέπει να μπορούν οι περιφέρειες να έχουν το δικαίωμα να διαλέγουν από, μη, από ένα φάσμα των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων αυτές που εξυπηρετούν καλύτερα τις τοπικές ανάγκες. Και αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μπορεί να επιλέγει περιφέρεια δύο-τρεις παρεμβάσεις, από τις πέντε ή έξι που είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Ανάλογα με τις ε, ανάγκες της, επαναλαμβάνω. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα ήθελα να σας καθησυχάσω, μην ανησυχείτε καθόλου. Πολλοί ζήτησαν το λόγο από την αίθουσα. Έχουμε ερωτήσει και από τις διπλανές αίθουσες και από το Twitter. Οι Ευρωπαίοι φιλελεύθεροι θεωρούν ότι το θέμα της ενέργειας θα πρέπει να μας απασχολήσει φέτος, δηλαδή να έχουμε παραγωγή η ενέργεια σε μικρή και μεσαία κλίμακα και να μειώσουμε τα ορυκτά καύσιμα, διότι πολλές ΜΜΕ και πολίτες ενδιαφέρονται για παραγωγή καθαρής ενέργειας. Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την μετάβαση, πώς μπορούμε να την προωθήσουμε. Δεν πρόκειται για μέσα. Δεν έχουμε πάντα τα πιο ε, ενισχυμένα μέσα Επίτροπε Χάνε, είπατε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε έργα υποδομής, αλλά δυστυχώς δεν έγιναν πάντα οι κατάλληλες επενδύσεις για τις ΜΜΕ από πλευράς ε, και καινοτομία και ούτω καθεξή. Θα ήθελα να, πω γιατί, να ρωτήσω γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς προτάσεις. Θεωρούμε ότι το 20% των ε, μέσων μας ε, χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Και ε, το ΕΤΠΑ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν τα καταφέρνει πάντα να εντάξει αυτό το 20% των δαπανών στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Και αυτό το 20% δεν ίσχυσε στο, στην περίπτωση του ΕΚΤ και του Ταμείου ε, Συνοχής. Ο κύριος Λάμπερτς, ευχαριστώ. Ακόμα και αν είναι επιτυχής η δέκατη αυτή εκδήλωσή μας, δεν πρέπει βεβαίως να ξεχνάμε πως δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Ευρώπη. Και αν θέλουμε να πάνε ξανά καλά τα πράγματα στην Ευρώπη, τότε δεν μπορούμε απλά να διαπιστώνουμε ε, ποιον φίλο πιανού πράγματος θέλουμε να ακούσουμε. Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα εάν καταφέρουμε οι άνθρωποι στη χωριά, στα καφενεία, στις περιφέρειες να πιστέψουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσθέμενη αξία. Και αυτό σχετίζεται με τις μεσοπρόθεσμες μεσονομικές προοπτικές. Γι' αυτό η δική μας η ομάδα θέλει να πει ξεκάθαρα πως υποστηρίζουμε τις προτάσεις της Κομισιόν και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για το ότι και το Κοινοβούλιο έχει την ίδια Αλλά τώρα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα γρήγορα και σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Και τέλος, πρέπει να υπάρξει μια εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Αυτό είναι παντού σημαντικό, αλλά σημαντικό είναι να μην διατρέξουμε τον κίνδυνο να μην υπάρχει πλέον η δυνατότητα επενδύσεων των ε, μορφών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμη προσκεκλημένη, θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για το κυρίως θέμα αυτών των ανοιχτών ημερών. Θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση όμως μεταξύ των διαφόρων θέσεων. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο προβληματικούς τομείς, στην ανεργία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Δυστυχώ έχουμε τεράστια έξαρση τη ανεργία ιδιαίτερα τη ανεργία των νέων. Και αν δεν κάνουμε κάτι θα χάσουμε ολόκληρε γενιέ. γιατί ε, χρέος των νέων να σπουδάζουν και χρέο δικό μα είναι να τους βρίσκουμε δουλειά μετά, να του εξασφαλίζουμε πρόσβαση στην αγορά εργασίας κάποια στιγμή θα τελειώσει η κρίση. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Και αυτό θα γίνει μόνο λύνοντας το πρόβλημα της ανεργίας, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων. Και με ανησυχεί η πορεία που πήραν το πρόγραμμα Έρασμος και άλλα προγράμματα. Έχει στο μυαλό της Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις για κινητικότητα των νέων. Επίση τι γίνεται με τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Είχαμε την συνεδρία στην Πολωνία και πολύ συχνά είχαμε κάποιες κεντρικές πρωτοβουλίες για την, ε, στη διάρκεια της κρίσης. Αλλά είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα που δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στην κεντρική διαχείριση, αλλά να αναγνωρίζουμε το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών, γιατί με συνεργασία μόνο μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικά πράσινες περιφέρειες και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελπίζω κυρία Χιούμπνερ να προστατεύσετε τους πυλώνας και τις βάσεις των διαρθρωτικών πολιτικών που είναι σημαντικές για τις περιφέρειες. Κάνω ό,τι μπορώ για να δώσω το λόγο σε όλους, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ευχαριστώ. Πραγματικά πολύ σφοδρή η συζήτηση. Θα ήθελα να πω το εξής. Μερικές φορές ε, ε, Φαίνεται να πανικοβαλόμαστε. Μιλάμε για την με τη μεγάλη σημασία που έχει η πολιτική συνοχή και αυτό είναι γνωστό γιατί είναι ε, σημαντικός ορός των περιφερειών και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της κάθε περιφέρειας. Αλλά εγώ έχω άλλη ερώτηση εδώ. Είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε ένα σταθερό πλαίσιο, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για να δημιουργήσουμε κίνητρα και να μην έχουμε συνέχεια απλώς ε, διορθώσεις ε, των ε, δημοσιονομικών πλαισίων. Θέλουμε σταθερό προγραμματισμό, σταθερό δημοσιονομικό πλαίσιο και στο μέτρο του δυνατού και ελαστικό. Να έχουμε αρκετή ευελιξία. Παρακαλώ, σύντομη, και εσείς είστε τελευταίος. Αγαπητοί συνάδελφοι, του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και η Επιτροπή των Περιφερειών, υποστήριξαν εξ αρχής μία κατηγορία περιφερειών υποκαθεστώς μετάβασης όπως είχε οριστεί. Τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν την ευθύνη. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο προπλησμός για τις υπομετάβαση περιφέρειες δεν σημαίνει αύξηση του γενικού προϋπολογισμού, ούτε μείωση του προϋπολογισμού των πιο μειονεκτουσών περιοχών. Θα πρέπει να είμαστε αποδοτικοί για αυτό το καθεστώς. Μιλάμε για ένα ΑΕΠ από 65 μέχρι 80% του μέσου κοινοτικού ΑΕΠ και θέλουμε να αναζωογονήσουμε τον κοινωνικό ιστό. Θα πρέπει να υπάρχει περιφερειακή συνοχή όπως ορίζει η συνθήκη και μιλάμε για 290 περιφέρειες. Δεν θα πρέπει να προβαίνουμε στο διαχωρισμό, ε, να αρκεστούμε στο διαχωρισμό φτωχές ή πλούσιες περιφέρειες. Θα πρέπει να καινοτομήσουμε. Πολύ σύντομα. Και μετά θα πρέπει να κλείσουμε. Ο συνάδελφος μίλησε για εδαφική συνοχή που σημαίνει χρηματοοικονομική προσπάθεια για να θεσπίσουμε αυτές τις ε, υπομετάβαση περιφέρειας. Υπάρχει όμως και μια άλλη προαπέτηση, συντονισμό της ΚΑΠ με την περιφερειακή πολιτική, διότι και η ΚΑΠ είναι παράγων συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και απασχόλησης. Δεν θα πρέπει να συγκλίνουμε τις προσπάθειες παρά να μιλάμε για ένα σύστημα όπου λέμε ισχύει ή η ΚΑΠ ή η συνοχή. Χρειαζόμαστε και τις δύο. Ευχαριστώ. Η πολιτική συνοχή, η διαρθρωτική πολιτική δεν είναι αυτοσκόπη. Πρέπει να συνεισφέρουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ευρώπη και σημαντική συνεισφορά σε αυτό είναι η πολιτική υγείας και η ευρωπαϊκή πολιτική βεβαίως έχει βάλει στις συνθήκες την αρχή της πολιτικής υγείας που θα πρέπει να σωματώνεται σε όλους τους άλλους τομείς πολιτικής. Κύριε Επίτροπε Χαν, πώς βλέπετε με όλες τις ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ κρατών, μελών και περιφερειών την ευθύνη της περιφερειακής πολιτικής για την πολιτική υγείας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήσασταν και σύντομοι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις, αλλά στις θέσουμε επιτάπητος. Θέλαμε τις ομάδες ε, και το Twitter. Το KGO ρωτάει κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης. Επίσης από, από το Ράντοσλαφ Ζαβάσκι από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιφερειακής ε, Συνεργασίας. Ποιος είναι ο ρόλος των ΜΚΟ μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας με τις βιομηχανίες, τους ακαδυναμικούς. Στο Twitter επίσης ο Κέβιν Ρος ε, μας ρωτά κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μείωση των ορυκτών καυσίμων και Υπάρχει μία άλλη ερώτηση από το Twitter από τη Σουηδία για την ε, ισότητα των δύο φύλων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο πάνελ. Μην απαντήσετε σε όλες τις επιμέρους ερωτήσεις, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Κύριε Πίτροπε, είπατε να ζει κανείς ή να μη ζει. Αν πρέπει να ορίσετε μία προτεραιότητα σε μία πρόταση έτσι ώστε να κρατήσουμε την αξιοπιστία μας, να κάνουν τη διαφορά οι περιφέρειες, ποια θα ήταν αυτή η πρόταση. Πρόεδρος και μετά ε, ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να δώσουμε αυτές απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Also die Regionalpolitik ist äh, das... Ναι. Η περιφερειακή πολιτική νομίζω είναι βασικό κομμάτι της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά την εφαρμογή τη συγκεκριμένη των διαφόρων στόχων. Όποιο πιστεύει λοιπόν στο όραμα της Ευρώπης χρειάζεται την περιφερειακή πολιτική και για την υγεία που αναφέρατε και σε αυτό μπορεί να συνεισφέρει η περιφερειακή πολιτική και από την πλευρά των υποδομών και από οποιαδήποτε άλλη πλευρά του ΙΣΕΦ e αλλά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αλλά έχουμε βεβαίως ε, και την προσέγγιση των πολλαπλών ταμείων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σας ευχαριστώ κύριε Χίμπνερ. Συγγνώμη, εγώ θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν συζητήσαμε και νομίζω είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ πέρα υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αποσταθεροποίησης της κατάστασης των περιφερειών που τώρα θα πρέπει να κάνουν και πολλέ επενδύσεις για να βγουν από την κρίση και νομίζω πως υπάρχει ο κίνδυνος πολλών διορθώσεων των προγραμμάτων λόγω της σύνδεσης με, τον ε, με τα εθνικά προγράμματα και τις ε, ε, εθνικές αυτές συστάσεις και τη γενικότερη μακροοικονομική κατάσταση. Οπότε δεν θα πρέπει να αποσταθεροποιήσουμε αυτή την πολιτική επενδύσεων και στο πλαίσιο αυτό και η μακροοικονομική αιρεσιμότητα και οι αλλαγέ που μπορεί να επιφέρει στι πληρωμέ και στις δεσμεύσει σε έργα που έχουν ξεκινήσει και είναι στη μέση θα έχει επίσης αποσταθεροποιητικό αποτελέσματα. Και ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με αυτά είναι αυτό το οποίο ανέφερε ο πρόεδρο Σούλτ. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα έλλειμμα μεταξύ 10 και 10 δισεκατομμυρίων που δεν βρίσκονται στον κοινοτικό προπολογισμό να πληρώσουμε λογαριασμού που έρχονται από τα κράτη-μέλη, από τι περιφέρειε και αφορούν έργα που έχουν ξεκινήσει οι δε διαχειριστικέ αρχές δεν θα έχουν λεφτά θα σταματήσουν τα έργα. Ε, αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί από το ότι προτείνουμε στο νέο πλαίσιο πολύ μικρές προκαταβολές λόγω της ε, δημοσιονομικής δε κατάστασης στο περιφερειακό και εθνικό επίπεδο θα μειωθούν τώρα και οι προκαταβολές στο 1% Οπότε όλοι αυτοί οι απλήρωτοι λογαριασμοί θα προσθεθούν στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές και υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος όπως είπα άρα για τη σταθερότητα της πολιτικής στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό με ανισχύει ιδιαίτερα. Μάλιστα. Άρα ας ευχαριστήσουμε τους ομιλητές. Αν υπάρχει ένα κεντρικό μήνυμα το οποίο απορρέει είναι ας προωθήσουμε την υπόθεσή μας. Θα πρέπει να έχουμε μία ενιαία και δυνατή φωνή και οι ανοιχτέ ημέρες αυτό ακριβώς προωθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, ζητώ συγγνώμη γιατί έπρεπε όλοι να είμαστε πειθαρχημένοι και θα ήθελα να σας καλέσω σε μία δεξίωση για, με βάση μία έκθεση από τις 6.30 μέχρι τις 8. Πρόκειται για μία έκθεση η οποία αφορά την διαπεριφερειακή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. vivía solamente de la agricultura. El gran colchón era la agricultura y ha desaparecido